Okay, you Ωραία. Τώρα θα καθυστερήσουμε, οπότε πρέπει να καθίσετε και να αρχίσουμε. Έγινε μια πολύ χρήσιμη και μεγάλη μακρά συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά λήφθησαν τόσο πολλές αποφάσεις που και ίδια έχω εκπλαγεί που τα καταφέραμε τόσο καλά, χάρη στην εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς των συναδέλφων. Και τώρα αρχίζουμε με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Στο έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 24ης Σεπτεμβρίου. Ορίστε κύριε Μαριά. Με τη γραμματεία, πολύ σύντομα, μίλησα προηγουμένως και με τη γραμματεία, να προσθεθεί στα minutes η πρόταση που είχαμε κάνει ο CCR για να υπάρξει δημόσια ακρόαση για το θέμα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων. Θα δούμε τις λεπτομέρειες με τη γραμματεία να προχωρήσουμε. Απλά σας το επισημαίνω αυτό για να καταχωρηθεί και θα τα δούμε αναλυτικά με τη γραμματεία. Ευχαριστώ. Excellent. Εξαιρετικά. Θα διορθωθούν δεόντως τα πρακτικά. Μάλιστα. Σημείο 4. Ανακοινώσεις δεν έχω ανακοινώσεις να σας κάνω, απλώς να ξέρετε ότι πήγα στον, στην Κύπρο <coughs> ως πρόεδρος της Επιτροπής μας <coughs> και η κάλυψη από τα μέσα ήταν και αυτή καταπληκτική, αλλά άλλο θέμα αυτό, άλλο άλλο. Τα διάφορα θέλει κανείς να προσθέσουμε τίποτα στην ημερησία διάταξη. Όχι. Τώρα για τους συντονιστές. Πήραμε πολλές αποφάσεις κάτι πολύ χρήσιμο για όλους μας για το μέλλον. Λοιπόν, εγκρίναμε, εγκρίναμε πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθώ εδώ τώρα να τα διαβάσω. Έχουμε εισηγητές. Θέλετε να διαβάσω όλα τα θέματα. Έχουμε την ετήσια έκθεση παραπραγμένων της Επιτροπής μας για το 2014 που θα αναλυφθεί από την Λιδία από τους σοσιαλιστάς και έχουμε εισηγητή για την ειδική έκθεση του διαμεσολαβητή, περί του διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού από κοινού με την ΛΥΜΠΕ θα είναι από το ΕΛΚ και θα συνεργαστεί με τον εισηγητή της ΛΥΜΠΕ. Για τις νομοδοτήσεις θα γίνει συντάκτης για την ετήσια έκθεση επιτήρησης ή εποπτεία τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 14 κάποιο από το ΕΛΚ. Και επίσης γνωμοδότηση προ την ΑΦΚΟ για την εφαρμογή της έκθεσης για τους Ευρωπαίους πολίτες, για την πρωτοβουλία των πολιτών. Εδώ μαλώνουν ακόμα οι συντηρητικοί με τους φιλελεύθερους, αλλά υποσχέθηκαν ότι θα τα βρουν σύμφωνα με το σύστημα DONT έχουν ίσους πόντους, έξι και η μεν και η δε. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε για τον κατάλογο 3 για τις απαράδεκτες αναφορές. Έγινε συζήτηση και γι' αυτού και από το Δεκέμβριο θα υποβληθεί επισήμως αυτός ο κατάλογος. Επίσης εγκρίναμε τη διαδικασία για την τροποποίηση συστάσεων μετά από πολύ χρήσιμη συζήτηση. Η ιστοσελίδα εγκρίθηκε επιτέλους και θα έχει μια δοκιμαστική περίοδο περίπου τρίμηνη που ταυτίζεται απλώς με την πρώτη φάση της εφαρμογής του. Κατά τα άλλα τα αναβάλαμε γιατί δεν προλαβαίνουμε. Κάτι κατεπήγον. Υπήρξε αίτηση κατεπήγοντος για τα παιδιά, το έθεσε το ΕΛΚ, για την προστασία των παιδών και για τις απαγωγές, για θέματα απαγωγών. Και είχαμε πει ότι πρέπει πάντοτε να ακολουθούμε την κατεπήγουσα διαδικασία όταν πρόκειται για παιδιά. Αυτά ήταν οι ανακοινώσει μου για τους συντονιστές. Είναι παρούσα εδώ και η Επιτροπή, η Κομισιόν και τώρα περνάμε στις αναφορές που θα συζητήσουμε με βάση τις γραπτές απαντήσεις της Κομισιόν ή άλλα έγγραφα. Για το 7 υπάρχει η αναφορά 0393 Και μήπως είναι παρόν εδώ ο Ντέιβιντ Πέτρι Μήπως ο κύριος Αλεχάνδρο Ντελκάμπο είναι παρόν. Ναι, πάρα πολύ καλά. Και ο κύριος Βάλκε και ο κύριος Τόμσον επίσης. Όχι. Δεν είναι ο κύριος Τόμσον. Αλλά οι άλλοι δύο καλώς ορίσατε. Πολύ καλώς ορίσατε μάλιστα. Ας αρχίσουμε με τον κύριο Βάλκε ή μήπω με τον κύριο Δελκάμπο Δελκάμπο, Δελκάμπο, Δελκάμπο, Δελκάμπο. Ορίστε. Καλημέρα. Είμαι Ισπανός, δικηγόρος και φοροτεχνικός στις νήσους Βαλαρίδες τα τελευταία 25 χρόνια και το Φεβρουάριο του 2013 Αποφάσισα να καταγγείλω τη χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί εισήγαγε υποχρέωση ενημέρωσης για περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που έχουν οι κάτοικοι της Ισπανίας στο εξωτερικό. Πρόκειται για το περίφημο μοντέλο 720. Θεωρώ ότι η υποχρέωση αυτή αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ισπανικό Σύνταγμα για πολλούς και διάφορους λόγους. Εδώ θα επικεντρωθώ σε ένα μόνο λόγο. Στην Ισπανία σήμερα τα μόνα εγκλήματα τα οποία δεν παραγράφονται ποτέ είναι γενοκτονία, τρομοκρατία και η κατοχή περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό για το οποία δεν έχει ενημερώσει ο υπόλογος βάσει του μοντέλου 720. Και μην νομίζετε ότι πρόκειται για μεγάλους απατεώνες, για ανθρώπους που είναι βοηθημένοι στη διαφθορά κτλ. Όχι, πρόκειται για πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες γιατί αρκεί να έχουν έναν μικρό τραπεζικό λογαριασμό πάνω από 50.000 ή ένα διαμερισματάκι στη Γερμανία ή στην Αγγλία, ε, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν το περίφημο μοντέλο 720. Και τι επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν υποβάλει κανείς το μοντέλο αυτό ή το κάνει εκπρόθεσμα. Υπάρχουν κυρώσεις 5.000 και 10.000 ευρώ το ελάχιστο. Αν κάποιος δηλαδή 60.000, λογαριασμό 60.000 δεν τον δηλώσει, έχει αυτά τα πρόστιμα. Και το χειρότερο είναι ότι μπορεί να υπολογίσει την αξία όλων αυτών των προσωπικών στοιχείων στο εξωτερικό, η Ισπανία, και να το θεωρήσει ότι πρόκειται για κέρδος που συγκεντρώθηκε το τελευταίο χρόνο που δεν έχει παραγραφεί. Η αξία λοιπόν των αγαθών αυτών φορολογείται ως κέρδος και το κράτος παίρνει 40 με 50% του ποσού αυτού. Και επιπλέον με προσάυξηση 150%. Στην Ισπανία παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια τα φορολογικά δικήματα. Όμως στην περίπτωση αυτή δεν παραγράφονται ποτέ. Θεωρείται αδίκημα τόσο σοβαρό που δεν παραγράφεται ποτέ. Ακόμα δηλαδή και αν αποδείξεις ότι τα έχεις αυτά τα αγαθά και πριν από 10-15 χρόνια, τίποτα είναι σαν να έχεις κάνει πολεμικό έγκλημα. Και μπορεί να υπάρξει και κατάσχεση των περιουσιακών αυτών στοιχείων στο εξωτερικό. Με τις διατάξεις αυτές λοιπόν ουσιαστικά παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Νομολογία η Ισπανία, γιατί υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λένε ότι χώρες ε, μέλη μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία, προκειμένου να παραγράψουν ένα δίκημα, αλλά εδώ πέρα η Ισπανία δεν το δεν παρατείνει την προθεσμία, δεν παραγράφεται ποτέ το αδίκημα αυτό. Και επειδή είμαι φοροτεχνικό και έχω συναντηθεί με πάρα πολλού ανθρώπους που ξέχασαν να υποβάλουν τη δήλωση αυτή, διαπιστώνω ότι εξαιτία αυτής της νέας φορολογικής υποχρέωσης που έχει πάρα πολύ σοβαρά πρόστιμα και που δεν παραγράφεται ποτέ, διαπιστώνω ότι πάρα πολλοί διστάζουν να κατασταθούν στην Ισπανία και άλλοι που κατοικούν στην Ισπανία ε, σκέφτονται να φύγουν όπου φύγει φύγει γιατί είναι σαφές ότι όσοι κατοικούν στην Ισπανία και έχουν επενδύσει στο εξωτερικό τιμωρούνται με τη διάταξη αυτή. Έτσι λοιπόν όπως είναι διατυπωμένη αυτή η διάταξη πιστεύω ότι παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο γιατί πρόκειται για εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων και κεφαλαίων. Συνεπώς πιστεύω ότι επήγει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ζητήσουν από την Ισπανία να προχωρήσει σε εξαιρέσεις ή να τροποποιήσει σημαντικά το, τη διάταξη αυτή. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Άντωνη Βάλκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Ονομάζομαι Άντωνη Βάλκε. Είμαι Βέλγος και Βρετανός υπήκος, δικηγόρος στον ε, νομικό σύλλογο του Δικηγό Σύλλογου του Βελγίου. Έχουμε μία οργάνωση, την ε, EU Rights Clinic, και ήρθαν σε επαφή μαζί μας η Ισπανική οργάνωση Αμπούσος Ουρμπανίστικος, που εκπροσωπεί κατοίκους στην Ισπανία οι οποίοι κατηγορούνται για παραβιάσεις. Και ήρθα σε επαφή μαζί μας επειδή διάφορα μέλη τους εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για τους κανόνες που ισχύουν σχετικά με την δήλωση περιουσιακών στοιχείων που έχουν κάτι και της Ισπανίας στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε και ο Αλεχάνδρο πριν από λίγο, οι κανόνες αυτοί πιστεύουμε εμείς ότι δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει διαφορετική μεταχείριση στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ισπανία και στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός της Ισπανίας. Γιατί η δήλωση αυτή 720 αφορά μόνο περιουσιακά στοιχεία που κατέχει κάποιος στο εξωτερικό. Συνεπώς υπάρχει διακριτική μεταχείριση μεταξύ αυτών που έχουν επενδύσει στην Ισπανία και αυτών που έχουν επενδύσει εκτό Ισπανίας. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει πάρα πολύ τον εκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν σήμερα στην Ισπανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει διάκριση στους κανόνες αυτούς, γιατί αν συγκρίνεται από τη μια μεριά τις κυρώσεις, αν κάποιος υποβάλλει καθυστερημένα δήλωση, την 720 που έχει να κάνει με τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό και τις κυρώσεις, τα πρόστιμα που επιβάλλονται στην περίπτωση που κάποιος υποβάλλει λανθασμένη δήλωση, βλέπετε ότι είναι πολύ υψηλότερα από αντίστοιχες κυρώσεις στην περίπτωση που πρόκειται για σπανικά περιουσιακά στοιχεία. το πρόστιμο δηλαδή για καθυστερημένη δήλωση 720 είναι 1500 ευρώ τουλάχιστον, ενώ 100 ευρώ αν υπάρξει καθυστέρηση για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ισπανία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δυσανάλογα έτσι πλήττονται οι Ευρωπαίοι πολίτες σε σχέση με τους Ισπανούς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στην Ισπανία και δεν είναι Ισπανοί είναι πιο πιθανό να έχουν περιουσιακά στοιχεία εκτός Ισπανίας από ότι οι ίδιοι οι Ισπανοί. Ιδίω θα δούμε πώς είναι οι συνταξιούχοι που ζουν στην Ισπανία. Επίσης πιστεύουμε ότι αποτελεί και περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την πλευρά του επανειλημμένως έχει πει ότι εθνικά μέτρα τα οποία δημιουργούν διακρίσεις ή εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου με το εξωτερικό, οδηγούν σε περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι οι κανόνες αυτοί εμποδίζουν και τις διασυνοριακές επενδύσεις. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν ένας Ισπανός κάτοικος στην Ισπανία θέλει να επενδύσει στο εξωτερικό αλλά καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσει πολύ παραπάνω για τις επενδύσεις αυτές στο εξωτερικό και κυρώσεις, προφανώς δεν θα το προτιμήσει, θα προτιμήσει επενδύσει στην Ισπανία. Υπάρχουν ε, και διάφορες υποχρεώσεις. Οι προθεσμίες είναι διαφορετικές όταν κάποιος έχει περιουσιακά στο εξωτερικό από ότι όταν έχει στο εσωτερικό. Υπάρχουν διαφορές. Μάιος Ιούνιος είναι η προθεσμία για τη δήλωση 720. Λάθος, λέει ο μιλητής. Τέλη Μαρτίου είναι η προθεσμία για το 720, ενώ για δηλώσει περιοριστικών στοιχείων στην Ισπανία είναι πολύ αργότερα. Αν ένα κάτοικο στην Ισπανία έχει επενδύσει στο Βέλγιο, έχει κάνει επενδύσει εκεί, τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλει για τις επενδύσεις αυτές θα δοθούν το Μάιο από, τις, από τα βελγικά αυτά ιδρύματα. Που είναι όμως πολύ αργά γιατί δεν προλαβαίνει να τα υποβάλει στη δήλωση 720 η οποία πρέπει να υποβληθεί πολύ νωρίτερα όπως είπαμε στην Ισπανία. Άρα εδώ υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση λοιπόν για τα ισπανικά περιουσιακά στοιχεία και εκείνα του εξωτερικού. Τι κάναμε εμείς. Κάναμε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητήσαμε από την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση και θα θέλαμε να δούμε να αλλάζουν οι κανόνες αυτοί. Να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και για την περίπτωση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και για περιουσιακά στοιχεία στην Ισπανία. Να υπάρχουν οι ίδιε προθεσμίες, τα ίδια πρόστιμα. Γιατί αν θέλουμε να εντοπίσουμε την φοροαποφυγή, πιστεύουμε ότι οι κανόνες αυτοί ξεπερνούν πολύ τα αναγκαία. Είναι δυσανάλογες οι διατάξει αυτέ γιατί καλύπτουν μόνο τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Γιατί αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη φοροαποφυγή, τότε θα πρέπει να ισχύει για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όχι μόνο για εκείνα που έχει ένα κάτοικος της Ισπανία στο εξωτερικό. Τέλος, έχει εκφραστεί ανησυχία για το πού πάνε οι δηλώσεις αυτές. Υπάρχουν διάφορε προτάσεις στην Ισπανία. Εξετάζουμε το να δημιουργηθεί ένα πράγμα που λέγεται exit tax, που σημαίνει ότι αν κάποιος δεν κατοικεί φορολογικά στην Ισπανία, να είναι υπόλογος σε ένα ειδικό ταμείο που έχει να κάνει με του, τα άτομα αυτά. Οι δηλώσει αυτές επίσης 720 φοβούμαστε ότι είναι μόνο η αρχή που θα οδηγήσει και σε άλλες άδικες μεταχειρήσεις και να οδηγεί σε περιορισμό των περιουσιακών στοιχείων των ατόμων αυτών στο εξωτερικό, μπορεί κάποια αρχή δηλαδή να πάρει τα χρήματα αυτά, κάποιο είδου κούρεμα. Για αυτού του λόγου λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να ερευνηθεί παρετέρω το θέμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Επιτροπή σα που δέχτηκε να εξετάσει την αναφορά μα αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε λάβει πολλές αναφορές για το θέμα αυτό. Είναι κάτι που αφορά και ενδιαφέρει πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Και δεν ήθελα να πω ότι η συζήτηση αυτή, η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Ξέρω ότι την παρακολουθείτε πολύ και θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς τα εσάς. Είμαστε η μόνη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κάνει απευθεία έκκληση στους πολίτες για να μας ενημερώσουν για τα θέματα που τους απασχολούν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Μαρία Λούιζα Τεβρίση και μετά θα υποβάλουν οι ευρωβουλευτές ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Λουίσα Τσίβρης και εκπροσωπώ την Κομισιόν σήμερα για τις τρεις αναφορές που συζητάτε. Αρχίζω με μια ενημέρωση. Στη κάτω την προκαταρκτική μας έρευνα, με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε, και θα προσπαθήσω να απαντήσω αργότερα και σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Σας επιβεβαιώνω ότι το θέμα το έχουμε εξετάσει όσο το δυνατόν σοβαρότερα. Οι αναφορές είναι για μας ένας πόρος πληροφόρησης για να γνωρίζουμε τι μπορεί να μην λειτουργεί σωστά στα κράτη-μέλη. Όπως σας είπαμε και γραπτός προηγουμένως, προσέξαμε ιδιαίτερα το θέμα ότι από το 2013 η Ισπανία έχει επιβάλει αυτή την ε, υποχρεωτική δήλωση περιουσιακών στοιχείων και στο εξωτερικό που επιβάλλεται και στους κατοίκους της Ισπανίας και στα άτομα και στις εταιρείες. Εφόσον οι φορολογούμενοι έχουν περιουσία και στο εξωτερικό. Κάναμε μια πρώτη έρευνα λοιπόν με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε. Ήρθαμε σε επαφές πολλές με, ισπανικές, με τις ισπανικές αρχές, συναντήσεις μέχρι και χθες είχαμε εκπρόσωπο των Ισπανικών Αρχών στο γραφείο μας για την περίπτωση αυτή. Ο διάλογος ήταν χρήσιμος, μας επέτρεψε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα στο μυαλό μας. Για να δούμε δηλαδή γιατί πρόσφατα εγκρίθηκε αυτό το νομοσχέδιο υποχρέωση. Δεν υπήρχε προηγούμενο ούτε για μας ούτε τις Ισπανικές αρχές. Δεν ξέραμε πώς θα εφαρμοζόταν ακριβώς αυτή η διάταξη, ποιες θα ήταν οι κυρώσεις ή γενικά οι επιπτώσεις εάν κάποιος δεν δήλωνε όπως έπρεπε τα περιουσιακά του στοιχεία. Και όπως λένε και οι αναφέροντες, τους οποίους ευχαριστούμε για όσες πληροφορίες μας έδωσαν, δεν επρόκειτο για θέμα που το έχουμε συνηθίσει στην περίπτωση αυτή είναι πολλές πτυχές χρειάστηκε να εξεταστούν, όχι μία όπως συνήθως σε φορολογικά θέματα. Και ασχολήθηκαν και πολλές υπηρεσίες της Κομισιόν. Γι' αυτό και η απάντησή μας ήταν κάπως μακροσκελής. Η διαδικασία κράτησε μάλλον πολύ χρόνο, αλλά πάντως οι αναφέροντες που είναι 40 με 50 μίλησαν για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και εμείς προσπαθήσαμε να δούμε επειδή υπάρχει πολύ μικρή εναρμόνιση για τα φορολογικά και είναι δικαιοδοσία των χωρών μελών βασικά πώς να φορολογήσουν και τι μέτρα να λάβουν, το μόνο που είναι υποχρεωμένο να κάνουν είναι να μην το κάνουν με διακριτική μεταχείριση. Ο στόχος του νομοσχεδίου φαίνεται να είναι η σωστή πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων των Ισπανών φορολογουμένων. Δηλώνοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία, ε, δίνουν μέσω στοιχεία και για τα ε, παρελθόντα εισοδήματά τους και για μελλοντικά εισοδήματα που μπορεί να πρέπει να φορολογηθούν στην Ισπανία. έγινε λόγος για το γιατί γίνεται λόγος ειδικά για περιουσία στο εξωτερικό και όχι στην Ισπανία, διότι για τα ισπανικά περιουσιακά στοιχεία έχουν περισσότερα μέσα στη διάθεσή τους οι αρχές για να διαπιστώσουν αν είναι πράγματι εκεί λογαριασμοί κτλ. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει για τα στοιχεία στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά το δικαστήριο στην ομολογία του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πει πολλές φορές ότι μπορεί να υπάρχουν θεμητοί λόγοι για τον περιορισμό ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως για φορολογικούς λόγους αλλά πρέπει να είναι αναλογική η περιορισμοί αυτή. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, οι υπηρεσίες της Κομισιόν έχουν αμφιβολίες ως προς τις επιπτώσεις που βγάζει το νομοσχέδιο αυτό για την καθυστερημένη υποβολή ή μη υποβολή των στοιχείων αυτών. Και τις αμφιβολίες αυτές τις εκφράσαμε και στις Ισπανικές αρχές. Και αυτή τη στιγμή αναμένουμε αν οι Ισπανικές αρχές δεν απαντήσουν μπορεί να συνεχίσουμε την έρευνα και περαιτέρω. Και επίσης επειδή η Κομισιόν στις σχέσεις της με τους αναφέροντες έχει αναλάβει την υποχρέωση να τους πληροφορεί τακτικά για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ετοιμάζουμε, έχουμε ήδη ετοιμάσει μία επιστολή όπου πληροφορούμε τους αναφέροντες για τα συμπεράσματά μας. Αυτή τη στιγμή μεταφράζεται γιατί πρέπει να απαντούμε στον αναφέροντες στη γλώσσα στην οποία μας απευθύνθηκαν, θα χρειαστούν ένα-δυο εβδομάδες ακόμα και θα λάβουν επομένως την ανάλυση μας, εκτεταμένη ανάλυση και θα έχουν και τη δυνατότητα να απαντήσουν μέσα σε ένα μήνα όπως συνηθίζεται. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα αλλά και η Κομισιόν έχει ωραία Είναι υποχρεωμένη μέσα σε 10 μέρες να κάνει μια πρώτη απάντηση στο Κοινοβούλιο για το πού βρίσκεται η αναφορά. Αν υπάρξει αλλαγή θα σας την υποβάλουμε γραπτός. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Αν υπάρχουν απορίες... Ωραία, αρχίζει η συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων. Πρώτα ο κύριος Μαρτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες για τα όσα μας είπαν, όπως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή λέει ότι απάντησε καλά η Ισπανία όσον αφορά αυτά τα θέματα και υπάρχει απόφαση για συνεργασία. Είναι πολύ βασικό. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ερευνούν. Αυτό είπε στο τέλος να έχουν περισσότερες πληροφορίες, να αναλύσουν λεπτομερώς και όταν θα τελειώσουν θα στείλουν στους αναφέροντες το αποτέλεσμά τους. Είναι καλό αυτό, είναι σωστό, οπότε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου φαίνεται λογική. Να τους δώσουμε ό,τι χρόνο χρειάζονται, δεν χρειάζεται να κλείσουμε τώρα την αναφορά αυτή, κάθε άλλο. Πρέπει να διευκρινιστεί τι είναι το καλύτερο. Αλλά δώστε μου και δύο λεπτά για να δούμε τι τελικά ζητάει ουσιαστικά αυτή η αναφορά. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε με την πρόθεση της νομοθεσίας να καταπολεμήσει την διαφθορά. Γιατί ορισμένοι μεταφέρουν τα περιουσιακά του στοιχεία στο εξωτερικό όλο και περισσότερο, όμως κάτι πρέπει να γίνεται γι' αυτό. Η δήλωση αυτή 706 αυτό θέλει ενημέρωση για να μπορεί να ελέγξει τα έσοδα των ε, ατόμων που είναι φορολογικά υπόλογοι στην Ισπανία. Ανεξάρτητα με το που βρίσκονται τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Νομίζω ότι είναι κάτι λογικό, θεμητό και όλοι συμφωνούμε για τον στόχο της νομοθεσίας αυτής. Το κατά πόσο κάνει διακρίσεις Φαίνεται πως όχι όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων και κεφαλαίων. Γιατί? Γιατί η ίδια η συνθήκη αναφέρει ότι χωρίς να προκαταλάβουμε κλπ. Και εδώ τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διατάξεις στο δικό τους φορολογικό σύστημα για να αντιμετωπίσει φορολογικά ο οποίους έχουν διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία σε διαφορετικά μέρη, λίγο πολύ. Άρα φαίνεται να μην υπάρχει διάκριση εδώ. Το ίδιο και όσον αφορά τις διευκολύνσεις. Γίνεται εύκολη η δήλωση αυτή. Όσον αφορά το, την παρέμβαση στον ιδιωτικό βίο το απόρριτο, δεν υπάρχει τέτοια διάκριση και τα στοιχεία τα οποία ζητάει η δήλωση αυτή για τα οικονομικά στοιχεία δεν αποτελεί τέτοια παραβίαση του απορρίτου γιατί είναι μέσα στα πλαίσια των μοντέλων που εφαρμόζονται και είναι γνωστά δεν παρεβιάζει το ιδιωτικό βίο. Συνεπώ χρειάζεται συνεργασία και να ξέρουμε ότι το γενικό συμφέρον είναι αυτό το οποίο πρέπει να υπερέχει. Όπως και να έχει το πράγμα, το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχουν περιορισμοί και διαφορές, ναι, αλλά να είναι αναλογικά όλα αυτά με το πρόβλημα. Έτσι όπως το βλέπουμε εμείς λοιπόν, υπάρχει αναλογικότητα αυτή των μέτρων δηλαδή που έχει οθετήσει η Ισπανική κυβέρνηση με αυτό που προσπαθεί να πετύχει. Ελπίζουμε ότι όταν έχουν τα τελικά του συμπεράσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή θα μας τα δώσει και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Μάτο. Πού δεν σε μπάγιο τώρα. Ναι, μάλιστα. Α, έχεις. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμηθεί η φορολογική αμπάτη, όμως με αυτά που ακούσαμε εδώ κατάστη σαφές το τι συμβαίνει στην Ισπανία, τι προσπαθεί να κάνει η Ισπανία. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά στους ε, πολιτικούς κύκλους της Ισπανίας, διαφθορά ευρύτατη και πιστεύω ότι η Ισπανία προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτήν την βαθιά διαφθορά. Και αυτό φυσικά δεν θα έπρεπε να αφορά τους ε, συνταξιούχους οι οποίοι έχουν εργαστεί όλη τους τη ζωή και αποφασίζουν να περάσουν ε, τα χρόνια της σύνταξής του στην Ισπανία. Φυσικά προσπαθούν λοιπόν να πιάσουν αυτούς τους φοροφυγάδες. Ωστόσο πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα καταφέρουν οι αρχές να εντοπίσουν αυτά τα διαφυγόντα κέρδη, πώς θα διαπιστώσουν σε ποιους ανήκουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και πώς σε περίπτωση που διαπιστωθούν αυτές οι παραβιάσεις, πώς θα επιστρέψουν τα χρήματα στο Ισπανικό κράτος. Φυσικά, να ε, επαναλάβω ότι οι ποινές είναι πάρα πολύ ψηλές στην Ισπανία για τις παραβιάσεις αυτές, ιδιαίτερα υψηλές, ασυνήθιστα υψηλές. Γενικότερα όμως η Ισπανία έχει πολύ αυστηρές ποινές και σε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα στις διαδηλώσεις. Ωστόσο, το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία αυτών των μέτρων. Είναι αυτά μέτρα τα οποία έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις ε, αργότερα και μιλάω για τους ε, συνταξίχους οι οποίοι διαμένουν στην Ισπανία, οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πληροφορηθούν καταλήλως και εγκαίρως για τα δικαιώματά τους, για τις ε, υποχρεώσεις τους και στις γλώσσες τους επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλα σχόλια ή άλλες ερωτήσεις. Σολεδάδ. Πρώτον, στην Ισπανία σήμερα ζούμε μια κατάσταση όπου το κράτος δικαίου το έχουμε χάσει, όπου η δικαιοσύνη και οι δυνάμεις του κράτους έχουν σαν ένα αποτέλεσμα να υπάρχει καταστολή και δίωξη. Δεν θα έλεγα ότι είναι διεφθαρμένη χώρα η Ισπανία. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι υπάρχει δίωξη της ε, διαφοράς. Είναι επίσης σημαντικό όμως να δούμε και το εξή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή. Όχι μόνο στην Ισπανία, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί και αλλού, γιατί φοροδιαφυγή υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε και κοινή αντιμετώπιση. Κατόπιν τούτου, για τη συγκεκριμένη αναφορά, δύο ζητήματα τίθεται. Το ένα είναι ουσίας και το άλλο είναι τύπου. Για το θέμα ουσίας, πιστεύω ότι είναι σαφές ότι τα άτομα τα οποία έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν για τα περιουσιακά τους στοιχεία, στο εξωτερικό είναι άτομα τα οποία είναι φορολογικά υπόλογα στην Ισπανία. Δεν πρέπει βέβαια να υπάρχει διπλή φορολόγηση, έτσι. Γιατί τότε θα ήταν άδικο. Επί της ουσίας λοιπόν φαίνεται ότι είναι ένα μέτρο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, λίγο πολύ κατά αναλογία. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είναι φορολογικά υπόλογα στην Ισπανία. Γι' αυτό έχουν αυτή την υποχρέωση. Τώρα, για το θέμα της διαδικασίας. Οι συνέπειες, τα πρόστιμα ή η διαδικασία μπορεί να είναι πράγματα τα οποία είναι δυσανάλογα ως προς τον ε, στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Επ' αυτού λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί πράγματι να συγκεντρώσει όσο περισσότερα στοιχεία μπορεί, να δει τι έχει μάθει από τις διάφορες φορολογικές και άλλες ισπανικές αρχές, να προχωρήσει τη διαδικασία και πιστεύω και εγώ πράγματι ότι πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία, αλλά επί της ουσίας το ζήτημα είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αυτός είναι ένας ευρωπαϊκός στόχος. Και αυτό πρέπει να δούμε και από πλευράς της Ισπανίας. Ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή διευκρίνηση. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις για το σε ποιον εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή. Δεν είναι νομοθεσία για του φτωχού Ευρωπαίου συνταξιούχου. Είναι μια νομοθεσία που αφορά όλου του φορολογικά υπόλογου στην Ισπανία. Και σε μένα. Και εγώ κάνω φορολογική δήλωση για τα περιουσιακά μου στοιχεία στις Βρυξέλλε. Και η συνάδελφο προφανώς και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι μόνο για του συνταξιούχου. Είναι για όλου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όλοι πληρώνουμε φόρους. Και στο σπίτι μας και εδώ. Θα ήθελα όμως τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντελκάμπο. Να είστε σύντομος παρακαλώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Δεν είναι ανάγκη, αλλά μπορείτε να προσθέσετε κάτι αν θέλετε. <laughs> Eh, είναι σαφές ότι ο στόχος της νέας αυτής υποχρέωσης είναι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ένα δυσανάλογο μέτρο και που δεν δικαιολογείται. Και γιατί είναι δυσανάλογο γιατί ένας είτε συνταξιούχος είτε όχι που κατοικεί στην Ισπανία, μια οικογένεια, τρία αδέρφια ή ένα ζευγάρι που έχει έναν τραπεζικό λογαριασμό στη Γερμανία με 60.000 ευρώ μόνο, 30.000 αντιστοιχούν στον καθέναν, έτσι, επειδή το συνολικό ποσό είναι πάνω από 50.000, ενώ στον καθένα αντιστοιχούν μόνο 30, πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση αυτή. Αν το ξεχάσουν μπορεί ο Ισπανικός νόμος να τους επιβάλλει 5.000 για τον καθένα, τελικά να φτάσει στις 20-25.000 συνολικά. Και μπορεί να υποθέσουν ότι το ποσό αυτό είναι ένα κέρδος, παρόλο που μπορεί να είναι αποταμιεύσεις, μπορεί να είναι ένα μικρό διαμέρισμα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δυσανάλογο το μέτρο. Έπειτα δεν κάνει διάκριση για το κατά πόσο τα περιουσιακά αυτά στοιχεία βρίσκονται σε έναν φορολογικό παράδεισο ή αν βρίσκονται στη Γερμανία, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στη Γερμανία, όπου κάθε χρόνο οι, οι γερμανικές φορολογικές αρχές ενημερώνουν την Ισπανία για τους ε, τόκους που έχουν από τα ποσά αυτά οι φορολογικά υπόλογοι. Αυτό σας λέω ότι δεν γίνεται διάκριση, είτε πρόκειται για ένα μικρό διαμερισματάκι στην Αγγλία, στη Γαλλία, είτε σε φορολογικούς παραδείσους, δεν γίνεται καμία Έπειτα, γιατί λέω ότι δεν δικαιολογείται η διάταξη αυτή. Γιατί ο κατάλληλο τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς τη φορολογική απάτη δεν πρέπει να φορτώνει με ε, διαδικασίες δύσκολες ή που κοστίζουν. Γιατί κοιτάξτε εμένα, κέρδος μου αποφέρει το να βοηθά τον κόσμο να κάνει τέτοιες δηλώσεις που είναι περίπλοκες. Παρ' όλα αυτά καταγγελώ τη χώρα μου γι' αυτό γιατί μπορεί σε κάποιον να στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα, γιατί έτσι και κάνει ένα μικρό λαθάκι θα του κοστίσει 10.000 ευρώ, οπότε προτιμά να πληρώνει φοροτεχνικούς. Γι' αυτό λέω ότι το καλύτερο είναι βάσει της οδηγίας για τι αποταμιεύσει και άλλα τέτοια μέσα, έτσι να καταπολεμηθεί η φορολογική αυτή απάτη, μέσω ενημέρωση, αμοιβέ ενημέρωση. Πρόεδρος, δεν θέλω να επεκταθούμε περισσότερο και να μας το ξανεξηγήσετε, απλώς μήπως έχετε κάποια απάντηση. Δεν είσαστε υποχρεωμένος να πάρετε το λόγο, αλλά αν το επιθυμείτε, παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τελικά το θέμα είναι, είναι δυσανάλογοι κανόνες αυτοί, ναι ή όχι. Δεν θα πω πάλι στα επιχειρήματα τα οποία σας παρουσίασα ήδη για τις κυρώσεις, τις προθεσμίες κτλ. Γιατί να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το αν τα περισσότερα στοιχεία βρίσκονται στην Ισπανία ή στο εξωτερικό. Τέλος, υπάρχουν κανόνες ευρωπαϊκοί που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και οι φορολογικές αρχές μπορούν να ενημερωθούν για αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει οδηγία του 2011 για αμοιβαία αρρωγή σε φορολογικά θέματα και οδηγία για τις αποταμιεύσεις που υποχρεώνει τις χώρες μέλη να δίνουν αυτά τα στοιχεία. Γιατί δεν φτάνουν αυτά. Αυτό ρωτάω. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσουμε για αυτό το θέμα. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ πολύ που παίρνετε τόσο σοβαρά αυτή την υπόθεση και μπαίνετε στην ουσία και έχετε αυτό τον εκτενή διάλογο που μας είπατε. Το εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος, να ξέρετε, εκ μέρου των Ευρωπαίων πολιτών. Είπατε επίση ότι θα στείλετε αντίγραφο της επιστολής, θα στείλετε καταρχήν επιστολή στον αναφέροντα μετά το διάλογο και σας παρακαλώ ένα αντίγραφο να το στείλετε και σε εμά στην Επιτροπή μας εδώ. Άκουσα από τους συναδέλφους ότι η πρόθεση είναι να μείνει η αναφορά αυτή ανοιχτή μέχρι να έχουμε περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επανέλθουμε σίγουρα. Είμαστε στο σωστό δρόμο πιστεύω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει σκληρά, οι Ισπανικές αρχές συμμετέχουν και μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι εδώ για να εξυπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. Και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο με διαφορετικά μέσα και δύο αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε και μας ενημερώσετε και να είσαστε σίγουροι ότι το θέμα σας θα το εξετάσουμε και πάλι μόλις έχουμε επόμενες πληροφορίες. Μπορείτε να παραμείνετε στην αίθουσα αν το επιθυμείτε ή να φύγετε όποτε θέλετε. Περνάμε στο επόμενο θέμα λοιπόν. Επόμενη αναφορά είναι η αναφορά 0967 του 2012. Έχουμε μαζί μας, ελπίζω, την Ζακλίν Κοτερίλ. Σωστά? Εδώ είσαστε. Ωραία, καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να στηρίξω τους ε, προηγούμενους αναφέροντας, διότι ως αντιδήμαρχος ε, στο χωριό μου στην Ισπανία καταλαβαίνω τα προβλήματα που υφίστανται. Η δική μου αναφορά αφορά το, τη στέρηση δικαιώματο ψήφου στου Ευρωπαίου πολίτε. Από καταρχά την Βρετανική κυβέρνηση, η οποία στερεί το δικαίωμα ψήφου στου Βρετανού πολίτε που ζουν στο εξωτερικό από 15 χρόνια και ε, πέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει στις ε, καταγγελίες και η Επίτροπος Ρέντιν έχει συμπεριλάβει το ζήτημα αυτό στην ε, ετήσια έκθεση για την Ιθαγένεια το 2014 και επικοινώνησε με τις ε, χώρες που μπλέκονται τον ε, Σεπτέμβριο. Η Βρετανική κυβέρνηση δήλωσε πως αν κερδίσει τις επόμενες εκλογές θα επεκτείνει το δικαίωμα ψήφου στους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό εφόρου ζωής. Αυτή ήταν μια καλή κίνηση, δεν ήταν όμως αρκετή. Χρειάζεται να αλλάξει η νομοθεσία έτσι ώστε να μας επιτραπεί να ψηφίσουμε στις, εθνικές, ε, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το αν η κυβέρνηση κερδίσει τις επόμενες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το θέμα είναι εάν η νομοθεσία θα τροποποιηθεί εγκαίρως. Το δικαίωμα εθνικής, ψήφου στις εθνικές εκλογές είναι αναφέρετο. Αυτή τη στιγμή εμείς ως Βρετανοί πολίτες δεν έχουμε το δικαίωμα ψήφου σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχουν και πολίτες άλλων χωρών οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές παρό... χώρα του τους παρότι διαμένουν σε αυτή. Όπως και εγώ, παρότι είμαι Μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου τη κοινότητά μου, δεν έχω το δικαίωμα ψήφου στι εθνικέ εκλογέ στην Ισπανία, ούτε στη Βρετανία. Τα τελευταία δέκα χρόνια λοιπόν δεν μπορώ να ψηφίσω και αυτό που είναι ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι έχω τρει ενήλικέ κόρε οι οποίε εργάζονται και πληρώνουν φόρου στην Ισπανία, δεν έχουν όμω το δικαίωμα ψήφου ούτε εκεί ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτή η δεύτερη γενιά μεταναστών εντό Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στερηθεί παντελώ το δικαίωμα ψήφου. Και αυτό είναι απαράδεκτο και συνιστά διάκριση εις βάρος της ηθαγένειας. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη ενίσχυσης των δημοκρατικών μας θεσμών και είναι ζωτική σημασία όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές και να είναι υπόλογες οι κυβερνήσεις απέναντί τους. Και είναι απαράδεκτο να μην μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης να ψηφίσει στη χώρα στην οποία εργάζεται και φορολογείται. Δεν πρέπει μόνο να έχουμε αυτό το δικαίωμα, πρέπει να έχουμε και το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στις χώρες στις οποίες διαμένουμε. Και να έχουμε το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στην ψήφο στη χώρα καταγωγής ή στη χώρα διαμονής. θα έπρεπε να δίδεται η δυνατότητα ψήφου σε πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό, έχουν όμως ε, διατηρήσει στενούς δεσμούς με την ε, χώρα καταγωγής τους. Σε μια έρευνα, πρόσφατη έρευνα, το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί πως πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα ψήφου σε πολίτες οι οποίοι διαμένουν επιμακρών σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει αποφανθεί ως εξή. Η αναγνώριση της στέρησης δικαιώματος ψήφου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό. Επίσης, προσθέτει ότι το Κοινοβούλιο έχει μέσα στη διάθεσή του έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσει και τα κρατημέλη και τα άλλα θεσμικά όργανα για ανάληψη δράσης. Ζητούμε λοιπόν, κάνουμε έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί για την έβρεση λύσης. Ο γιος μου είναι 18 χρονών, θα γίνει μάλλον σύντομα 18 χρονών και όπως και πάρα πολλοί άλλοι θέλει να έχει το δικαίωμα να ψηφίσει και να μην θεωρείται πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Και ελπίζω να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει αυτό το βασικό δημοκρατικό του δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας κάνατε την εισαγωγή σε αυτό το σημαντικό θέμα. Τώρα η κυρία Κέρτεν Ντόλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω την αναφορά και την καμπάνια που έγινε σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο για την επέκταση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των βασικών δικαιωμάτων της ελευθερίας κυκλοφορίας ας πούμε που είναι μεγάλο θέμα που αφορά και την έξοδο από την κρίση, την κινητικότητα των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά όμως που συζητιούνται όλο και περισσότερο, τα δημοκρατικά δικαιώματα δεν συνοδεύουν αυτά τα δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μερικές χώρες όπως και η δική μου έχουν θέσει χρονικά όρια για την εφαρμογή των δημοκρατικών δικαιωμάτων όπως της ψήφου. Αν κανείς λείπει από το Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από 15 χρόνια χάνει το δικαίωμα να ψηφίζει σε βρετανικές εκλογές. Αυτό καταδικάζουν μεταξύ άλλων οι αναφέροντες και τα χρονικά αυτά όρια δηλαδή. Και το ίδιο ισχύει και για τις άλλες χώρες που έχουν θέσει τέτοιο χρονικό περιορισμό στην άσκηση δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Άκουσα ότι το κυβερνών κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο στο μελλοντικό του μανιφέστο υπόσχεται να καταργήσει αυτά τα όρια. Γιατί όμως δεν το κάνουν τώρα που είναι στην εξουσία, να ρωτιέμαι. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι υπάρχει δημόσια υποστήριξη για αυτό το αίτημα. Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και συμπολίτε μου δεν πιστεύουν ότι είναι σωστός αυτός ο περιορισμός των δικαιωμάτων. Και στην νομική επιτροπή έχουμε θέσει το θέμα και έχουν γίνει και άλλες δράσεις σχετικώς και γι' αυτό υποστηρίζω του, τις προτάσεις των αναφερόντων. Ωραία. Τώρα ζητώ συγγνώμη από την Κομισιόν γιατί είναι παρούσα αλλά δεν της έδωσα το λόγο. Έπρεπε να το είχα κάνει αμέσως μετά την παρουσίαση της αναφοράς. Τι Μπορμπάση λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για αυτό το πρόβλημα του υστέρησης δικαιώματος ψήφου και είναι ενήμερη από το 2013. Ανακοινώσαμε τότε ότι πρέπει να ληφθεί δράση για το ζήτημα αυτό, διότι πραγματικά υπάρχουν πέντε κράτη-μέλη στα οποία πολίτες που έχουν ασκήσει το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση χάνουν το βασικό δικαίωμα ψήφου. Αυτό λοιπόν ήταν, ένα, ήταν το πρώτο βήμα και φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μία σύσταση στα αντίστοιχα κράτη-μέλη, όπου αναφέρεται ότι αυτή η πολιτική στέρηση ψήφου στην ουσία τιμωρεί πολίτες που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ορισμένε επικοδομητικέ λύσει, όπω για παράδειγμα η έκκληση στα κράτη-μέλη να δώσουν τη δυνατότητα στου πολίτε τους να κρατήσουν, να διατηρήσουν το δικαίωμα ψήφου, εφόσον συνεχίζουν να επιδεικνύουν ένα συνεχές ενδιαφέρον για τα πολιτικά τεκτενόμενα της χώρας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ζήτησε από τα κράτη-μέλη αυτά να μην αφαιρούν αυτόματα το δικαίωμα ψήφου από τους πολίτες τους, αλλά όσοι πολίτες επιθυμούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας καταγωγής τους και το δείξουν αυτό το ενδιαφέρον να έχουν το δικαίωμα αυτής της συμμετοχής με την ψήφο στις εθνικές εκλογές. Και στη σύσταση αυτή συμπεριλήφθηκαν ορισμένα πρακτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν. Για παράδειγμα, προτείναμε υποχρέωση ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους πολίτες που διαμένουν στην Αλλοδαπή να είναι δυνατή και ηλεκτρονικά. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, πολίτες που διαμένουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος μπορούν να ε, ζητήσουν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις εθνικές ε, αυστριακές εκλογές. Αυτή λοιπόν είναι μια καλή πρακτική και εμείς ενθαρρύναμε τα ε, πέντε αυτά κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα όπως ε, της Αυστρίας. Και επίσης να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες και εγκαίρως για τις ε, προϋποθέσεις άσκησης αυτού του δικαιώματος ψήφου σε εθνικές εκλογές. Με αυτή τη σύσταση λοιπόν, με αυτό το σημαντικό έγγραφο που εκδόθηκε νωρίτερα το 2014, προσπαθούμε να οδηγήσουμε σε μία αλλαγή προς το καλύτερο. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως πραγματικά χαιρόμαστε με το ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται μια δημόσια διαβούλευση και μάλιστα με αφορμή τις τελευταίες εκλογές το θέμα αυτό ακούστηκε περισσότερο. Θεωρούμε πως αυτή η σύσταση ήταν μια ισορροπημένη προσέγγιση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι εθνικές εκλογές αποτελούν εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εκείνα είναι λοιπόν ε, νομικά αρμόδια να αποφασίσουν ποιο έχει το δικαίωμα να ψηφίζει στι εθνικέ εκλογέ. Τονίσαμε όμω ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βασικό θεμελιώδε δικαίωμα των ε, Ευρωπαίων πολιτών, την ελευθερία της μετακίνησης και πως αυτό δεν πρέπει να ε, αποκλεί την ψήφο σε εθνικές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την περιεκτική απάντηση. Θα συνεχίσουμε τώρα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζαμπόρσκα. Ζντανόκα, με συγχωρείτε λέει πρόεδρος. Ναι, ναι, τα σλαβικά ονόματα είναι δύσκολα για σας, τέλος πάντων. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που διατύπωσαν το αίτημά τους. Γιατί με την αναφορά αυτή βοηθάτε και μερικούς ευρωβουλευτές στον αγώνα για τα ευρωπαϊκά πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Δυστυχώς οι περισσότεροι εδώ μέσα, τουλάχιστον από την προηγούμενη θητεία το είδα, δεν θεωρούν ότι χρειάζεται τέτοια στήριξη. Και εγώ είχα κάνει μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ όπου ζητούσαμε η ευρωπαϊκή ηθαγένεια να θεωρείται σαν κάποια πρόσθετη αξία και να χορηγούνται δικαιώματα και στους Ευρωπαίους πολίτες που να μην απορρέουν αυτόματα και μόνον από τα δικαιώματα που έχουν ως εθνικοί πολίτες. Ιδιαίτερα στο θέμα <coughs> της συμμετοχής σε εκλογές. Δυστυχώς οι μισοί ευρωβουλευτές, λίγο παραπάνω από τους μισούς μάλλον, διαφωνούσαν. <coughs> σε μια άλλη έκθεση για την Ιθαγένεια όπου ζητούσε περισσότερα δικαιώματα για τους Ευρωπαίους πολίτες που να μην απορρέουν μόνο αποκλειστικά από τα δικαιώματά τους ως πολίτες κρατών πάλι απέτυχε. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η ισορροπία των δυνάμεων στο νέο κοινοβούλιο αλλά πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε. Γιατί το 2013 ήταν το έτος της Ιθαγένειας και όλες οι εκθέσεις των διαφόρων επιτροπών και ιδίως στην Επιτροπή Αναφορών έγινε λόγος μόνο για την ελευθερία της διακίνησης. Το μόνο δικαίωμα που αντιμετωπίσαμε, που συζητήσαμε ήταν αυτό. Τίποτε άλλο. Το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές όμως είναι πολύ σημαντικό και συμφωνώ ότι η περίπτωσή σας που εδώ είναι τρομερή για εσάς και τα παιδιά σας. Θα ήθελα λοιπόν, Πρόεδρε, να δούμε μήπως δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε κάποιο κείμενο για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ως Επιτροπή Αναφορών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τα εκλογικά δικαιώματα με βάση αυτή την αναφορά. Κάτι άλλο η Επιτροπή ανέφερε πέντε χώρες μέλη που παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το πρωτόκολλο 1, αν θυμάμαι καλά, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να οργανώνουν δημοκρατικές εκλογές και άρα να συμμετέχουν σε αυτές και όλοι οι πολίτες και εκλέγει και εκλέγεστε. Θεωρητικά λοιπόν θα μπορούσατε κυρία αναφέρουσα να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσετε να εξαντλήσετε όλα τα ένδικα μέσα εθνικά και είναι πολύ μακρά η διαδικασία. Αλλά είναι μια δυνατότητα. Τώρα επειδή θέλουμε και εμείς και το Συμβούλιο της Ευρώπης να εμφανιζόμαστε ως πρωταθλητές της δημοκρατίας πρέπει να υποστηρίξουμε και αυτή την αναφορά προφανώς. Ευχαριστούμε κυρία Σντανόκα. Καλά το είπα τώρα. Λοιπόν, και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέκερ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και στο όνομα της πολιτικής μου ομάδας, ε, του ΕΛΚ, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αναφέρουσα για την αναφορά αυτή, διότι πραγματικά μας δίνει την δυνατότητα να δείξουμε τη, την δύναμη αυτής της ε, Επιτροπής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και πιστεύω πως ε, η σύσταση αυτή πρέπει να μας κάνει να ασχοληθούμε με το ποια είναι τα όρια της επικουρικότητας. Διότι εδώ υπάρχει μία αντίφαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο, μία ε, δίκαιο, μία αντίφαση ανάμεσα στο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, της ελεύθερης εγκατάστασης, το να μπορεί ο καθένας να πάει όπου θέλει και να κατοικήσει όπου θέλει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη να χάνεται ένα ακόμα θεμελιώδης δικαίωμα, το δικαίωμα ψήφου το οποίο είναι βασικότατο θεμελιώδες δικαίωμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 στην έκθεση για τα δικαιώματα των πολιτών αναφέρει ότι είναι αναφέρεται και πλήρες δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να συμμετέχουν ενεργά ως Ευρωπαίοι πολίτες στις εκλογικές διαδικασίες και η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα κράτη αυτά καθιστά σαφή παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Γι' αυτό λοιπόν, προτού εμείς ως Επιτροπή αναλάβουμε δράση, θα ήθελα να προτείνω να διεξάγουμε μία ακρόαση στην Επιτροπή Αύκο Συνταγματικών Υποθέσεων. Υπάρχει δυνατότητα τον ε, Δεκέμβριο και στην ακρόαση αυτή της ΑΦΚΟ μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς, να ασχοληθούμε με αυτό ακριβώς το θέμα και μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αυτήν την αναφορά και μετά να εξάγουμε και τα συμπεράσματά μας προτού δραστηριοποιηθούμε ως Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεμπάγιος. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ για την θετική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι πραγματικά προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στα κράτη-μέλη όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου. Στη Σουηδία συζητούμε εδώ και καιρό για μία αλλαγή της νομοθεσίας περί ηθαγένειας και πραγματικά ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα για διπλή ηθαγένεια και ένα επιχείρημα εναντίον τη διπλή ηθαγένεια είναι ακριβώ αυτό, το να έχει κάποιο το δικαίωμα ψήφου σε δύο χώρε. Εμεί όμω θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται από το ότι υπάρχει πολύ μικρή συμμετοχή στις εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται περισσότερη ενεργή, ενεργό συμμετοχή στις εκλογές, περισσότερο ενδιαφέρον στην πολιτική και αυτό δεν θα γίνει τόσο εύκολα. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μένουν σε μια χώρα και καταγόνται από κάποια άλλη και θέλουν να ψηφίσουν εκεί. Πραγματικά, ε, λέει η Πρόεδρος, ε, με αυτά που κάνετε μας κάνετε περήφανος που είμαστε Σουηδοί. Μπέατρις, έχετε το λόγο τώρα. Δεν με έχετε συνηθίσει να μιλώ Σουηδικά, έτσι. Αλλά και εγώ πρέπει να το θυμάμαι μερικές φορές ότι είμαι Σουηδέζα. Ναι, μα μιλάτε τόσο πολλές γλώσσες, σας ζηλεύω πραγματικά. Εγώ θα μιλήσω ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα θέλω να πω για την αναφορά αυτή. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Κοτερίλ και γιατί μας έφερε την αναφορά αυτή που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τους λόγους που θα σας εξηγήσω αλλά και επειδή αποτελεί παράδειγμα για το ότι λειτουργεί, κάνει τη δουλειά της η Επιτροπή Αναφορών. Το 2006 λοιπόν η κυρία Κατριλάλ μας έφερε μία αναφορά για να σταματήσει ένα οικοδομικό σχέδιο για το Αλικάντε. Και όντω, είναι ένα παράδειγμα για το ότι η Ευρωπαϊκή Αναφορών λειτουργεί για πράγματα σημαντικά, συγκεκριμένα και για την πρωτοβουλία των πολιτών. Το δεύτερο για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κοτερίλη είναι γιατί Παίρνει ένα θέμα εδώ, το οποίο πέρα από τις νομικές διαστάσεις που έχει και πώς εμπλέκεται σε αυτά ακόμα και η Συνταγματική Επιτροπή, θέτει και πάλι το θέμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, το δικαίωμα ψήφου δηλαδή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει άμεση σχέση με την έννοια της Ιθαγένειας. Το κατά πόσο λοιπόν πρέπει κανείς να δείχνει τη σχέση που έχει με τον χώρο στον οποίο ζει ή αν αρκεί να είναι κανείς Ευρωπαίος πολίτης. Εγώ στηρίζω λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή απόλυτα και όπως και με την ομάδα μου έχουμε το Let Me Vote που ισχύει από το 2011 για τις ευρωεκλογές αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε ότι εξετάζονται επιλογές. Επιπλέον όμως θέλω να κάνω έκκληση. Να λάβουμε υπόψη μας ότι οι νέοι που είναι το μέλλον της Ευρώπης και που είναι σε τόσο δύσκολη κατάσταση σήμερα όσον αφορά το μέλλον τους πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να είναι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες και άρα να μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μίτση έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω μια σπανία γλώσσα. Μαλτέζικα. Και θέλω να σας πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τις θέσεις όλων και της κυρίας Κοταρέλ πρώτα απ' όλα η οποία βάζει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και μπορώ να καταλάβω την απογοήτευσή της και εκείνη της οικογένειάς της. Ζει σε μια άλλη χώρα, συνεισφέρει, αλλά περιορίζονται τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να ψηφίσει στη χώρα αυτή. Καταλαβαίνω λοιπόν την απογοήτευσή της. Αντιλαμβάνομαι και την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε τι έχει γίνει για το θέμα. Αλλά πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί. Γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για μια περίπτωση που έχει μια λύση για όλους. Και θα σας πω γιατί. Εγώ προέρχομαι από μια μικρή χώρα, την Μάλτα, 400.000 κάτοικοι, και στις κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα μου, 230.000 πάνε και ψηφίζουν στις εκλογές. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί Μαλτέζοι, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν όλοι αυτοί οι Μαλτέζοι που ζουν στο εξωτερικό ψήφιζαν για μια κυβέρνηση στην Μάλτα, στην οποία όμως δεν ζουν. Καταλαβαίνετε ότι και εδώ τίθεται ένα θέμα δημοκρατίας και ελεύθερης διακίνησης. Ελπίζω ειλικρινά να βρούμε μια λύση για όλες τις χώρες. Συνεπώς η Επιτροπή με αυτά που είπε στο τέλος να παραμείνει στα πλαίσια των τοπικών κυβερνήσεων, των εθνικών κυβερνήσεων. Οι ανάγκες, θέλω να πω, χωρών όπως η Γερμανία και η Ισπανία δεν είναι ίδιες με εκείνες άλλων μικρών χώρων, όπου κινδυνεύει να υπάρξει κάποια ανισορροπία. Συνεπώς, η λύση που θα πρέπει να βρούμε πρέπει να είναι μία λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε χώρας χωρίς βέβαια να εμποδίζουμε τη δημοκρατία, αλλά συγχρόνως σεβόμενοι τα δικαιώματα όλων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανάγκες μερικές φορές διαφέρουν και αποκλίνουν. Οι μικρές χώρες δηλαδή δεν πρέπει να θεωρηθούν αλλιώς. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, αλλά η άσκηση του δικαιώματος αυτού συνάδει με κάποιες ευθύνες. Εύχομαι λοιπόν ότι καλύτερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πετύχει μια λύση σεβόμενη την ισορροπία αυτή και να υπάρχει η καλύτερη λύση για τις ανάγκες της κάθε χώρας. Η κυβέρνηση, είτε περιφερειακή είτε εθνική της κάθε χώρας έχει τελικά την ευθύνη. Ο κύριος τώρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. συζητούμε για θέματα που είναι πολύ ευαίσθητα στις χώρες μας. Όταν μιλάμε για το δικαίωμα ψήφου, μιλάμε και για το δικαίωμα στην εθνικότητα της κάθε χώρας και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια συγχρόνως. Μια που ο καθένας μας έχει διπλή ηθαγένεια. Μια εθνική, η υπηκότητα που έχει δηλαδή, και επιπλέον έχει και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αν καταλαβαίνω καλά την αναφορά που μας υποβάλλεται από Βρετανή πίκο η οποία κατοικεί στην Ισπανία επιμονή μου βάσεως, το εμπόδιο για αυτήν είναι διπλό. Γιατί επειδή ζει πάνω από 15 χρόνια εκτός Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές της χώρας της, του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί συνεπώς να εκλέξει αυτούς που εκπροσωπούν τους πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γαλλία έχουμε κάτι αντίστοιχο, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με τη διάρκεια διαμονής στο εξωτερικό. Απλώς και μόνο με το γεγονός ότι κάποιος διαμένει στο εξωτερικό. Κάποιος που δεν έχει διεύθυνση στη γαλλική επικρότεια δεν μπορεί να ψηφίσει για τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Και στις τελευταίες εθνικές εκλογές το 2012 προσπαθήσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και τι κάναμε, είπαμε ότι θα υπάρξουν κάποιοι εκπρόσωποι των ομογενών, των Γάλλων δηλαδή που ζουν στο εξωτερικό. Η Γαλλία πάντα θεωρεί τον εαυτό της ε, έτσι, παγκόσμιο. Οπότε χωρίσαμε τον κόσμο σε 11 επικράτειες ένας Γάλλος που εδώ και ένα, δύο, 15, 30, 40 χρόνια ζει στην Αυστραλία, εκπροσωπείται από έναν βουλευτή της περιοχής Ασία και Ειρηνικός, ο οποίος εδρεύει στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Είναι ένας Γάλλος, ο οποίος ψήφισε για έναν Γάλλο βουλευτή που τον εκπροσωπεί. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα της αναφοράς με το οποίο συμφωνώ. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο που λέει ότι αν κατοικούμε σε μια χώρα τις οποίες δεν έχουμε την υπηκότητα, παρόλα αυτά θα ήταν λογικό εκτός από τις τοπικές εκλογές να μπορούμε να ψηφίζουμε και για το Εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας αυτής. ξεχνάμε ότι οι βουλευτές αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι τροποποιούν και το σύνταγμα της χώρας. Ε, στη Γαλλία διαφωνήσαμε γι' αυτό. Ένας Ευρωπαίος δηλαδή πολίτης, ο οποίος κατοικεί στη Γαλλία, μπορεί να ψηφίσει στις τοπικές εκλογές, Μπορεί και να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, αλλά δεν μπορεί να είναι δήμαρχος γιατί αυτό συνδέεται με τους γερουσιαστές και τίθεται θέμα κυριαρχίας. Κάποιοι συνάδελφοι λένε όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, θα έπρεπε όλοι να μπορούμε να ψηφίζουμε. Ναι, είμαστε όλοι Ευρωπαίοι πολίτες. Στις ευρωπαϊκές εκλογές μόνο οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών ψηφίζουν όπου και αν κατοικούν, ναι, αλλά είναι ευρωπαίοι πολίτες. Οι άλλοι πολίτες οι οποίοι κατοικούν στις χώρες μας, αλλά που δεν έχουν την υπηκότητα κάποιες από τις 28 χώρες, δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές. Με αυτή τη γραμμή λοιπόν πρέπει να ευθυγραμμιστούμε κι εμείς και να προσέχουμε να μην βάλουμε στο τραπέζι κάτι το οποίο τελικά θα οδηγήσει στο να επανέλθει ο κόσμος στο δικαίωμα της υπηκότητας και μόνο. Κινδυνεύουμε έτσι να ενισχύσουμε το αίσθημα το αντιευρωπαϊκό ορισμένων συναδέρφων ή και ορισμένων ε, πολιτών χωρών που δεν έχουν φεντεραλιστική προσέγγιση. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύει ότι δεν πρέπει να πάμε πιο μακριά. Σας είπα ότι από το αντικείμενο της αναφοράς διαφωνώ με ένα τμήμα και συμφωνώ με ένα άλλο τμήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα, κύριε Κοτερέλ, θέλετε να πάρετε και πάλι το λόγο για τελευταίες παρατηρήσεις, παρακαλώ. Ναι. Ε, θα είμαι σύντομη γιατί περνάει ο χρόνος, το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Ευρωβουλευτές και την Επιτροπή σας για την σημερινή σας στήριξη στην ανηφορά. Δεν πρέπει να τιμωρούμε κάποιον επειδή θέλει να σκίσει το δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία. Όντως έχουμε μια γενιά οι οποίοι κυκλοφορούν στην Ευρώπη ψάχνοντας δουλειά και που φεύγουν από τις χώρες τους για 5, για 10 χρόνια ή και για παραπάνω. Θα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν εκεί όπου ζουν και εργάζονται. Το γεγονός ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Τζούρι στήριξαν ε, το θέμα της ψηφοφορίας στη χώρα στην οποία κατοικεί κανείς σημαίνει ότι αυτό είναι εφικτό εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα καθεστώ όπου θα έχουν τα ίδια δικαιώματα όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε όπου και αν κατοικούν. Ελπίζω ότι η Επιτροπή σα θα συνεχίσει να στηρίζει την αναφορά αυτή, να την εξετάζει και να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα πριν περάσουν πολλά χρόνια. Για κάτι που ακούσαμε από την κυρία Μπεθέρα για την προηγούμενη αναφορά που υπέβαλα εδώ, όντως άλλαξε τα πράγματα. Ελπίζω ότι και αυτή τη φορά θα κάνετε πολύ καλή δουλειά και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τα καλά αποτελέσματα αυτά σύντομα. Όπως καταλάβατε όλοι ενδιαφέρονται για το θέμα σας. Εγώ καταλαβαίνω την αντίδραση της Επιτροπής. Όλοι θεωρούν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και δεν θα το λησμονήσουν. Και τώρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Άκουσα να λένε οι συνάδελφοι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Εγώ θα ήθελα να καλέσουμε τον κύριο Τίμερμανς ως αρμόδιο αντιπρόεδρο για θέματα της Επιτροπής μας να έρθει να μας δει για να εξετάσουμε το θέμα. Η αρμοδιότητά του είναι βελτίωση της νομοθεσίας και μας είπε στην ακρόασή του ότι θα έρθει στην Επιτροπή μας όσο το δυνατόν συντομότερο. Να μια χρυσή ευκαιρία να τον καλέσουμε για να συζητήσει το θέμα μαζί μας. Θα το προτείνω αυτό και ίσως να πούμε και στην Κομισιόν ότι να επανέλθει και αυτή για να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συμβαίνει στις πέντε χώρες που αναφέρατε. Ποιες είναι οι πέντε χώρες. Και μετά προτείνω επίσης ως Επιτροπή Αναφορών να γράψουμε και επιστολή στην, σε προσώπους της Βρετανικής κυβέρνησης, του υπεύθυνους, του αρμόδιους και να τονίσουμε τη σημασία που έχουν τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Συμφωνείτε, μάλιστα ευχαριστούμε πολύ. Πάει και αυτό το θέμα, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Κυρία Κοτερίλ, Μπορείτε να παραμείνετε αν θέλετε, αλλά μπορείτε και να φύγετε. Τώρα η αναφορά 9, το σημείο 9 για τις δημόσιες προμήθειες του Φούλβιου Αλμπάνων και άλλων για την παραβίαση της οδηγίας 2004 κάθετος 18 της Κομισιόν για τις δημόσιες συμβάσεις. Και η κυρία Λούρα Βέσα είναι παρούσα μάλιστα. Θα δώσω το λόγο αμέσως σε εσά. Σας ευχαριστώ. Η αναφορά υποβλήθηκε από μια οργάνωση παραγωγών ιατρικού υλικού σε άμεση σχέση με τις δημόσιες αγορές και προμήθειες Η οδηγία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναδιαπραγματεύονται το ύψος των συμβολέων των συμβάσεων. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις πρακτικά διότι οι οργανισμοί που ασχολούνται με την υγεία δεν αρκούνται στην αναδιαπραγμάτευση του ύψους των ποσών αλλά και στις ίδιες τις ρήτρε των συμβολέων και των συμβάσεων. Συζητήσαμε λοιπόν με εκπροσώπους της διοίκησης της κυβέρνησης και για το ίδιο το περιεχόμενο της σύμβασης του συμβολέου και έγινε αναδιαπραγμάτευση των τιμών αναφοράς. Θέσαμε το ερώτημα στην Ιταλική κυβέρνηση που δημοσίευσε μία εγκύκλιο με το περιεχόμενο της συμφωνίας. Η κατάσταση όμως παραμένει δύσκολη. Ο νομοθέτης επανέλαβε ότι υπάρχει αυτή η αρχή της αναδιαπραγμάτευσης. Επειδή λοιπόν μειώθηκαν κατά 5% τα ύψη των συμβάσεων των συμβολέων αναδιαπραγματεύτηκαν και το περιεχόμενο της ίδιας της Ρήτρε χωρίς καμία εξήγηση από την Ιταλική κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις μας επομένως πρέπει να αναδιαπραγματευτούν συμβόλαια σε έναν τομέα για τον οποίο η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων είναι πολύ ψηλή η αναδιαπραγμάτευση των τιμών έχει σαφείς επιπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων, στην ποσότητα των προϊόντων που περνάνε από τις δημόσιες αγορές και προμήθειες και όλα αυτά παραβιάζουν μάλλον την οδηγία 18 του 2004 για τις δημόσιες αγορές και προμήθειες που προβλέπει απαγόρευση της αναδιαπραγμάτευσης και σεβασμό του ανταγωνισμού. Απαγορεύει τις προσφορές που είναι περιέργως χαμηλές και η Ιταλική κυβέρνηση επομένως πρέπει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα γιατί αλλοιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών που χορηγούνται στους πολίτες έτσι. Σίλβιο Γρήγο, εκ μέρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την αναφέροντα. Ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το 2012, από εκεί ξεκίνησε. Ο ίδιος ο κανόνας του 2012 έχει να κάνει με παραβίαση των ε, κανόνων των δημοσίων ε, προμηθειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Μάρκτα πιο συγκεκριμένα, ήρθαν σε επαφή με τις ταλικές αρχές προκειμένου να τεθούν οι ερωτήσεις που έπρεπε να τεθούν και για να αποσαφινιστεί η ερμηνεία του κανόνα γιατί πράγματι θα μπορούσε να υπάρξει παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες. Γι' αυτό καθόλου τη διάρκεια εγκυρότητας της σύμβασης. Το κύριο πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής. Ο κανόνας αποκλεί πολύ συγκεκριμένα την ε, δυνατότητα τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης. Μπορεί να τροποποιηθεί η τιμή υπέρ της υγειονομικής αρχής σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν θα μπορούσε να τροποποιηθεί η διάρκεια της σύμβασης. Δεν υπήρχε όμως καμία απαγόρευση για την τροποποίηση άλλων στοιχείων της σύμβασης. Και ακριβώς εδώ είναι που υπάρχει πρόβλημα ερμηνείας. Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε διευκρινήσεις από τις Ιταλικές αρχές. Δημοσιεύθηκαν δύο εγκύκλοι από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών και η τελευταία εγκύκλιος είναι της 1 η Σεπτεμβρίου. Ίσως οι αναφέρουσαν να μην έλαβε γνώση της τελευταίας αυτής εγκύκλιου. Πάντω, σύμφωνα με τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εγκύκλιος αυτή εξηγεί και αποσαφηνίζει τους ορισμούς, τη δυνατότητα δηλαδή διαπραγμάτευσης για τα άλλα στοιχεία της σύμβασης. Η εγκύκλειος αυτή εξηγεί την δυνατότητα διαπραγμάτευσης που δεν μπορεί να έχει σαν στόχο παρά μόνο την τιμή και όχι τα άλλα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης. Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλειο αυτή, οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν ότι το θέμα όσον αφορά την ερμηνεία διευθετείται. Και οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισαν να μην αρχίσουν να μην μπουν στη διαδικασία επί παραβάση που θα ήταν το επόμενο στάδιο. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εγκύκλειος αυτή μας βοηθάει να αποφύγουμε μια διοικητική διαδικασία που θα παραβίαζε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η δυνατότητα, δυνατότητα δηλαδή τροποποίησης των ουσιαδών στοιχείων. Θέλει κανείς το λόγο παρακαλώ. Πίτερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην αναφορά αυτή έχουμε ταυτόχρονα και καλά και κακά νέα. Από τη μία καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν διατάξεις οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να διαλευκανθεί το ζήτημα. Και μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για οικονομικά συμφέροντα εδώ στις συμβάσεις αυτές. Υπάρχει όμως από την άλλη και το θέμα της ε, υγείας, ο τομέας της υγείας και δυστυχώς εδώ είναι δυσάρεστο το ότι χρειάζονται ακριβώς ε, δύο χρόνια μέχρι να δούμε τι γίνεται νομικά και να διασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια δικαίου. Το καλό από την άλλη είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και και υπάρχει μια συμφωνία όσον αφορά την ε, νομική βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε μια εγκύκλιο που κυκλοφόρησε, όμως ε, δεν την, έλαβε, δεν την έλαβαν οι αναφέροντες. Και υπάρχει εδώ πέρα ένα πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα στην ε, κυβέρνηση της Ιταλίας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι βλέπω. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους αναφέροντες. Αυτή η εγκύκλειος σας είναι γνωστή. Τη λάβατε. Εντάξει, αν μου πείτε όχι, τότε τελείωσε. Αλλά εάν την έχετε λάβει, εάν σας είναι γνωστή. Η εγκύκλειος αυτή έλυσε τα βασικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην αναφορά σας. Και εάν δεν έφτασε η εγκύκλειος, τότε θα ήθελα να προτείνω να παρακολουθήσουμε στενά την κατάσταση και να ζητήσουμε από τους αναφέροντες να ε, παραμείνουν σε επικοινωνία μαζί μας και να μας ενημερώσουν για τα νεότερα. Τώρα, θα ήθελα να απευθυνθώ στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους εμπλεκόμενους και να τους ζητήσω να επιληθούν όσο το δυνατόν συντομότερα αυτά τα οικονομικής φύσης προβλήματα τα οποία έχουν ε, διαπιστωθεί εδώ. Διότι πραγματικά εάν επιμείνουν αυτά τα προβλήματα θα είναι ένα ακόμα λιθαράκι προς όφελος των ευρωσκεπτικιστών. Γι' αυτό λοιπόν συνοψίζοντας υπάρχουν και καλά νέα και κακά νέα με αυτήν την αναφορά. Ευχαριστώ Πίτερ. Άλλος? Κανείς. Η αναφέρουσα λοιπόν έχει το λόγο. Όχι, εμείς δεν ενημερωθήκαμε για την εγκύκλιο αυτή. Υπάρχει ο νέος νόμος το 2014, μετά από δύο χρόνια δηλαδή, που επιβεβαιώνει την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης χωρίς να αναφέρει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο, όπως δηλαδή και το 2012. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε για την εγκύκλιο αυτή. Καμία υγειονομική αρχή από αυτές με τις οποίες είμαστε σε επαφή δεν μας ενημέρωσε, δεν μας έδωσε κανένα στοιχείο για την εγκύκλιο αυτή. Οπότε η κατάσταση παραμένει ίδια για μας. Πίτερ. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αναφορά διότι έτσι καλλιώς πιστεύω πως μία εγκύκλειος δεν είναι απόρριτο έγγραφο και θα ήθελα να το λάβει η αναφέρουσα ή αναφέροντας. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμεσολαβήσει και να του το διαβιβάσει, διότι είναι πραγματικά βασικό. Εκείνοι, όσοι, εκείνοι που έχουν ε, επηρεαστεί από το θέμα αυτό να είναι και ενημερωμένοι μέσω της εγκυκλίου. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Μια απλή αποσαφήνιση, Πρόεδρε. Έλαβε πληροφόρηση 18 Αυγούστου κατέσσερα η αναφέρουσα από την Κομισιόν όπου τις λέγαμε ότι οι Ιταλικές αρχές ήταν έτοιμες να εγκρίνουν την εγκύκλιο. τι το είπαμε αυτό. Όπως είπε και η ίδια στην αρχή της παρέμβασής της. Και εμείς λάβαμε λοιπόν την εγκύκλιο αρχές Σεπτεμβρίου και στη μελλοντική μας απάντηση θα το αναφέραμε που είναι δημόσιο έγγραφο φυσικά και άμα θέλει να της δώσουμε το κείμενο και τώρα. Ωραία. Αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί. Όσο δεν έχει αποσαφινιστεί θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Σωστά. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και οι υγειονομικέ αρχές να λάβουν γνώση της ε, κυκλίου. Γιατί αν και οι ίδιε δεν γνωρίζουν την ύπαρξή της, τότε δεν προχωράμε πουθενά καθόλου. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα η Κολίν Μπαϊνές έχει το λόγο. 6.47 αναφορά του Colin Blinders, βρετανική Σταγέννη, εξ τη της Corporative Group, Greenpeace κλπ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Colin Baines. Ή Colin Baines. Ή. Α, όχι, δεν είμαι η Colin Baines. η α οχι δεν ειμαι colin baines προσωπώ μια οργάνωση μεταφορών που έχει συνυπογράψει αυτή την αναφορά σας είχα στείλει μία παρουσίαση Bauer δεν ξέρω αν τη λάβατε. Με διαφάνειες, με απ' όλα. Πού είναι? so that we are now just taking a Α, ναι, μάλιστα. Ψάχνουμε την παρουσίαση των διαφανειών, μάλιστα. Έχουμε το μηχάνημα, έχουμε, έχουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Okay, so Ωραία. Δεν ξέραμε καν αν ήσασταν παρούσα στην αίθουσα, τέλος πάντων. Η εκπρόσωπος των αναφερόντων λοιπόν έχει το λόγο. Με συγχωρείτε για την σύγχυση, αλλά δεν είμαι η Colin Baines, ο Colin Baines, το είπα και στην αρχή εκπροσωπώ τον Colin Baines όμως, γιατί η οργάνωσή μου έχει υπογράψει την αναφορά. Την αναφορά. Την αναφορά. Την αναφορά. Ωραία. Θεώρησα ότι καλύτερο θα ήταν να παρουσιάσω και μερικές διαφάνειες γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Η αναφορά υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2011 και συνοδευόταν από 15.000 υπογραφές και με από μια έκθεση εδώ έξω από το κοινοβούλιο στηρίζεται όπως σας είπα από το Cooperative UK που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων και τη δική μου οργάνωση καθώς και το WWF. Ζητάει βασικά από την Κομισιόν να εφαρμόσει μέτρα μείωση των πομπών αερίου θερμοκηπίου, με εφέ θερμοκηπίου. Θα σας εξηγήσω τι είναι η ασφαλτόδη Βλέπετε εδώ την εικόνα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Α, βλέπετε, α, καλά. Και θεωρείται το μεγαλύτερο βιομηχανικό σχέδιο παγκοσμίως. προς στιγμή η ασφαλτόδης άμμος μόνο στον Καναδά εξορίζεται, στην Αλμπέρτα. Αλλά τα σχέδια υπάρχουν και σε πολλές άλλες χώρες, Μαδαγασκάρη, Ρωσία, Νιγηρία κλπ. Τι είναι η οδηγία ποιότητος καυσίμων, είναι τμήμα μέρος της κλιματολογικής δέσμης που εγκρίθηκε το 9 με συγκεκριμένους στόχους για το 20. υποτίθεται στοχεύει στην δημιουργία καθαρότερων καυσίμων. Έχει ως στόχο 6% μείωσης των εκπομπών διοξιδίου και είναι το μόνο τμήμα του, της κλιματολογικής δέσμης που πέντε χρόνια αργότερα δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί όταν συζητιέται ήδη το καινούργια δέσμη. Έγινε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί το 11, η Κομισιόν δηλαδή πρότεινε ορισμένα εφαρμοστικά μέτρα τα οποία είχαν διαφορετικές τιμές, πρόβλεπαν διαφορετικές τιμές για τις εταιρείες. Η πρόταση εκείνη εφάρμοζε αυτά που ζητούσε ο αναφέρον από την Κομισιόν να κάνει να μειωθούν οι εκπομπές και να υποχρώνονται οι εταιρείε να αναφέρουν τι κάνουν. Τις ασφαλτόδεις άμμος τις θεωρούσαν σαν περίπου ισοδύναμες με το υγρό αέριο, το υγραέριο. Και γι' αυτό εφάρμοσαν διαφορετικές τιμές για το υλικό αυτό γιατί χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια για τη μεταποίησή του και την διήλυσή του είναι βασικά χειρότερο για το περιβάλλον από τα άλλα. Εδώ είναι στοιχεία μιας μελέτης της Κομισιόν που αποδεικνύουν ότι οι ασφαλτόδεις άμοι χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για να μεταποιηθούν. Και μετά το 2011 έγινε μια ψηφοφορία χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση για προβλήματα επιτροπολογίας. Και αυτό σημαίνει ότι επανήλθε η πρόταση στην Κομισιόν η οποία αποφάσισε να κάνει μια αξιολογική μελέτη η οποία υποστήριζε την αρχική πρόταση. Το 2014 όμως, δυόμιση χρόνια μετά, η Κομισιόν αποφάσισε να παρατήσει κάθε μέτρο για τα μη συμβατικά πετρέλαια ή καύσιμα έγιναν, ασκήθηκαν πιέσεις από τον Καναδά, τις Ηνωμένε Πολιτείε και τις πετρελαϊκές εταιρείες. Αν θέλετε τα στοιχεία τα έχουμε και λόγω των πιέσεων αυτών και των λόμπι υποχρεώνονται οι εταιρείε να αναφέρουν μόνο μία μέση τιμή εκπομπών των προϊόντων τους. Τι άλλαξε λοιπόν με την πρόταση του 14. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα. Το 11 δεν είχαμε συζητήσει τα στοιχεία, αλλά η πρόταση του 14 δεν υποχρεώνει πια τις εταιρείε να αναφέρουν τα στοιχεία για τα μη συμβατικά καύσιμα. Αν και υπάρχουν διαφορές στα είδη καυσίμων που χρησιμοποιούνται, θεωρούνται όλα ισότιμα ως προς τις εκπομπές. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος αντέδρασε σε αυτούς τους νέους κανόνες και ζήτησε εξηγήσει. Το χειρότερο είναι ότι η Κομισιόν μονομερός αποφάσισε να μην εφαρμόζει πια μετά το 20 του στόχους της οδηγίας. Και άρα δεν είναι πολύ στεναροί οι συνοδευτικοί κανόνες για την εφαρμογή της. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, καμία διαβούλευση με το κοινοβούλιο και επομένως στην ουσία δεν θα εφαρμόζεται καθόλου η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα και ελπίζω το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να θέτει το θέμα. Η, τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι πρέπει τα δύο τρίτα των ορυκτών καυσίμων να μην τα εξορίσουμε πλέον αν δεν θέλουμε να υπάρξει η σφαιρική θέρμανση που φοβόμαστε. Και για να γίνει αυτό θα έπρεπε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μη συμβατικά καύσιμα και να αρχίσει να συμμορφώνεται και η πετρελαιοβιομηχανία με τους στόχους των εκπομπών. Βέβαια, διεθνώ τα πράγματα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση και θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι οι 15.000 υπογράφοντες ζητούσαν κάτι που δεν έχει ακόμα γίνει, δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ή έχουν βάλει νερό στο κρασί τους. Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων είναι πολύ ζωτική για την κλιματολογική πολιτική και το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστεί διαφανής διαδικασία για τη λήψη ή μη της απόφασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ο Όιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μαζί μας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την αναφέρουσα που μας έκανε αυτήν την εισαγωγή και την παρουσίαση. Θα ήθελα να σας εξηγήσω σε ποιο στάδιο εφαρμογής της νομοθεσίας βρισκόμαστε. Όπως είπε και η αναφέρουσα, ήταν μέρος του πακέτου για το κλίμα το 2008-2009 και δυστυχώς μας πήρε πάρα πολύ καιρό για να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε. Αυτή τη στιγμή Βρισκόμαστε σε μια θέση όπου απέτυχε η διαδικασία επιτροπολογίας και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει κάποια πρόταση στο Συμβούλιο, το οποίο θα την συζητήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 6 Οκτωβρίου αυτή την πρόταση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα εξέτασης και απόφασης μετά. Υπήρξε μια συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος χθες και σημείωσα ότι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες συμφώνησαν να λάβουν ξεκάθαρη θέση για το θέμα αυτό. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί με πλειοψηφία να απορρίψει ή να εγκρίνει την πρόταση. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην διαδικασία. Καταρχάς αποφασίζει το Συμβούλιο προς τα που θα πορευτούμε και μετά το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα εξέτασης και έγκρισης ή απόρριψης της πρότασης. Η αναφέρουσα ανέφερε κάποια σημαντικά στοιχεία. Καταρχάς τις τιμές για την ασφαλτούχο άμμο. Υπάρχουν αυτές οι τιμές στη σελίδα 9 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι γεγονός. Πράγματι δεν ε, υπάρχει διαφοροποίηση ως πρώτη ύλη, αλλά ως ε, τύπος ε, καυσίμων. Όμως υπάρχει συμφωνία με το στόχο της μείωσης του 6%. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να γνωρίζει το ενεργειακό αποτύπωμα, το αποτύπωμα άνθρακα όλου του αργού πετρελίου που κυκλοφορεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και στις σελίδες 12 έως 15 μπορούμε να δούμε τις τιμές για τον Καναδά, στις σελίδες 30 έω 34 τις τιμές για τη Βενεζουέλα, η οποία είναι μία από τις χώρε που παράγουν αυτήν την ύλη από ασφαλή του χώμου. Πιστεύουμε πως αυτή η πρόταση είναι μια βελτίωση σε σχέση με το 2012-2013, διότι αυτή τη στιγμή εμείς ζητούμε την επεξεργασία όλης της γκάμας του αργού πετρελαίου, ενώ πριν γινόταν λόγος μόνο για συμβατικό ή μη συμβατικό πετρέλαιο. Τώρα όμως ζητούμε να μάθουμε τι ακριβώς εισάγεται, πόσο πετρέλαιο εισάγεται, από πού κτλ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για μια μελλοντική πολιτική. Η αναφέρουσα επίσης μίλησε για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σταματήσει ε, ε την προώθηση της ε, οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων από το 2020 και μετά. Ε, πράγματι, τον Ιανουάριο υπήρχε ένα σχετικό έγγραφο και είχαμε και, τις, ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου πριν από 10 περίπου μέρες όπου δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν και η απόφαση του Συμβουλίου οι οποίες δεν αναφέρονται σε κάποια συνέχιση της οδηγίας αυτής. Όμως με το που έχουμε περισσότερες γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό και μετά από την ε, σχετική διαβούλευση για την ε, συνολική μείωση κατά 40% θα ξέρουμε περισσότερα και θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τώρα όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα που πρέπει να μείνουν στο υπέδαφος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Πρέπει να βρούμε όμως και τρόπους να μειώσουμε γενικότερα τη χρήση ορυκτών καυσίμων και αυτό θα γίνει βελτιώνοντας την, ε, αποδοτικότητα και εξοικονομώντας πόρους γενικότερα. Πρέπει να βρούμε διαφορετικές λύσεις και διαφορετικούς τρόπους από το να χρησιμοποιούμε μόνο την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, διότι αυτή η οδηγία στόχο έχει να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα για τα καύσιμα προορίζονται για τις μεταφορές. Δεν έχει ως στόχο να ασχοληθεί με τις πρώτες ύλες, αλλά αυτό που σας είπα μέχρι τώρα και μέχρι το 2020. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές και η Μαργκρέτε να έχει το λόγο και μπορεί να αρχίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω δανέζικα. Όπως και εσύ μιλάς σουηδικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το... την αναφέρουσα. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί. Και εδώ δεν έχετε όποιον και όποιον. Πρέπει να ξέρετε ότι το περιβάλλον είναι αυτό που θέλουμε να έχει ένα σημαντικό ρόλο παντού. Και το θέμα λοιπόν που εξετάζουμε σήμερα είναι ένα από αυτά τα μικρά πραγματάκια που βοηθούν σε αυτό. Παρά λοιπόν τα επιστημονικά δεδομένα που γνωρίζουμε όσον αφορά τις ασφαλτούχες άμμους, λέμε ότι πρέπει να τοποθετηθούμε σαν να είναι ίδιο όπως και όλα τα υπόλοιπα. Στο θέμα των υδρογονοθράκων υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση και είναι ζωτική σημασία στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας, τα Εθνικά Κοινοβούλια, να κάνουμε τα πάντα ώστε το περιβάλλον να ξαναγίνει μια σημαντική υπόθεση για όλους και να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Η πράσινη ανάπτυξη είναι το στίχημα. Αν θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε παλιά, με επιδοτήσεις, με επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζονται, επιχορηγούνται κλπ, θα χάσουμε. Γιατί δεν θα πληρώσει το λογαριασμό μόνο το κλίμα, μόνο η φύση, αλλά και οι βιομηχανίες και η ευρωπαϊκή απασχόληση. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο για όλους. Δεν πρέπει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί όπως κάναμε μέχρι τώρα. Δεν πρέπει να τα κρύβουμε. Αντίθετα, πρέπει να τα προβάλλουμε. Τότε θα έχουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που να φανεί τι λέει. Αν πούνε δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, να ξέρουμε με ποια βάση το κάνει αυτό. Και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορεί να κρύβει τα προβλήματα. Αυτή πρέπει να είναι η θέση μας πιστεύω. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαστικαμά έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Χάζεκάμπ. Κάθε φορά που βλέπω αυτή την εικόνα, σοκάρομαι, πραγματικά όπως και με το σχιστολιθικό αέριο. Και με εκπλήσει που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει σαν στόχο το να απαγορεύσει του τα στέρεα ορυκτά. Αν δείτε τα δεδομένα και σκεφτείτε τις επιπτώσεις, το μόνο που μπορείτε να πείτε είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι. Συμφωνώ με το συμπέρασμα της συναδέρφου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λιγάκι έτσι στεύκολα ξεπετάει το θέμα όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Να τις μειώσουμε και τελειώσαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την έκθεση για το κλίμα και εκεί φαίνεται ότι τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε με τα στέρεα ορυκτά. Να αλλάξει η κατάσταση. Δεν έχουμε επιλογή, ούτε χρόνο στη διάθεσή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να κάνει περισσότερα ώστε να δώσει συνέχεια στην αναφορά αυτή. Ευχαριστούμε. Έχουμε άλλα 10 λεπτά. Έτσι, ε, πολυτέλεια στην Επιτροπή μας. Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Α, ο κύριος Μαντά, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κανένας ειδικό όσον αφορά τα ορυκτά, ούτε και ακόμα λιγότερο για την ασφαλτούχα άμμο. Ξέρω όμως ότι οι ασφαλτούχες άμμοι ρηπαίνουν πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην λαμβάνουμε υπόψη τους προσανατολισμούς μας για την επόμενη περίοδο που είναι η μείωση 40% εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια στην βιομηχανική στρατηγική που αντιβαίνει τελικά στους στόχους μας. Εγώ συμφωνώ να περιμένουμε λίγο. Εντάξει, είμαι μερικές φορές αφελής, ίσως γι' αυτό ξεκίνησε και με την πολιτική. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα 300 δισεκατομμύρια που μας υποσχέθηκε ο Γιούγκερ, μπας και υπάρχει εκεί μέσα κάποια ευχάριστη έκπληξη και κάποια δισεκατομμύρια πάνε ως επένδυση για την βιώσιμη ανάπτυξη της ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν η ιδέα είναι χρειαζόμαστε κι άλλο πετρέλαιο, οπότε μην κάνουμε τίποτα, συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα, τότε ειλικρινά φοβάμαι πάρα πολύ για τον πλανήτη μας. Ευχαριστώ λοιπόν που μας ενημερώσατε για αυτά, για να ξέρουμε τι συμβαίνει, γιατί μερικές φορές δεν ξέρουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά πάνω στον πλανήτη μας. Εγώ συμφωνώ ότι βιώσιμη ενέργεια θα έχουμε με βιώσιμες πηγές ενέργειας και θα έχουμε και απασχόληση, θα σώσουμε και τον πλανήτη και όπως λέω πάντα και το επαναλαμβάνω και τώρα, μας έχει εκλέξει ο κόσμος. Δεν ξέρω και τι λόμπι υπάρχουν από δίπλα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε μια τέτοια κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ. Ωραία. Προσπαθώ βασικά να ζητήσω τη βοήθειά σας, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν ε, τους αναφέροντες που μας ενημέρωσαν. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα προσπαθώντας να λύσει το ζήτημα αυτό. Δεν τα καταφέρατε γιατί είναι δύσκολο. Αλλά δεδομένου ότι και το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια δεν τα έχει καταφέρει καλά. Καλά θα κάνουμε και εμείς να είμαστε ταπεινόφρονες και να μην καταδικάζουμε τους άλλους αφού εμείς δεν τα καταφέραμε. Αλλά αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τώρα, και γι' αυτό ήθελα να πάρουν περισσότεροι το λόγο για να καταλάβω λίγο πολύ τι θέλετε, πώς θέλετε να συνεχίσουμε. Κανείς όμως δεν είπε αυτό θα ήθελα να κάνουμε. Οπότε, εγώ προτείνω να μείνει ανοιχτή αναφορά αυτή, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να το εξετάζει, να δει πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Δεδομένου ότι είχαμε και το πάνελ για το κλίμα και πολλές συναντήσεις, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε βοηθήσει έτσι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξάλλου έχουμε και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με νέες πολιτικές ιδέες ελπίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να επανέλθετε παρακαλώ με περισσότερο πολιτικό βάρος θα έλεγα στην απάντησή σας. Το άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να πάμε στην ΕΝΒΗ, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να τους ρωτήσουμε εκείνους τι προτείνουν. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά μπορούμε να απευθυνθούμε σε άλλες αρμόδιες επιτροπές και να του ζητήσουμε τη γνώμη τους. Συμφωνείτε να προχωρήσουμε έτσι, αν συμφωνούν οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές, το ΕΛΚ και εγώ. Γιατί δεν είμαι καθόλου ειδική στο θέμα. Αλλά τώρα νιώθω σαν να είμαι λιγάκι. Ωραία. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή όρεξη. Θα επανέλθουμε ανανεωμένοι μετά το γεύμα.